Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων. Περνώ απευθεία στο υπαριθμό ένα σημείο με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης και σας ενημερώνω για τις εξή αλλαγές στην ημερήσια διάταξη 9.34 34 και 56 είναι τα σημεία που αναβάλλονται. 51 είναι το σημείο το οποίο θα συζητηθεί μετά το 28. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις, θεωρείται εγκριθήσα η ημερήσια διάταξη με τις τροποποιήσεις αυτές και θα ήθελα να σας ενημερώσω πώς προβλέπετε μετάδοση από το διαδίκτυο για το θέμα αυτό, εκτός από τα σημεία της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και κλεισμένων των θυρών. Είναι δε ενδεικτικό απόλυτο στο χρονοδιάγραμμα και μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της συνεδριάζεως. Ανακοινώσει του Προέδρου, ε, σας ενημερώνω για τις αποφάσεις των συντονιστών της συνεδριάσεως της 24ης ε, Σεπτεμβρίου, όπου οι συντονιστές αποφάσισαν τον διορισμό των εξή εισηγητών. Του κύριου Γκράντε, Γκράντε Πασκουάλ για την έκθεση για την συμπληρωματική προστασία, το πιστοποιητικό συμπληρωματική προστασία. Το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασία για τα ιατρικά προϊόντα του κυρίου Κοφεράτη για την έκθεση για την ε, επίδοση στα κράτη-μέλη ε, εγγράφων σχετικά με, σχετικών με εμπορικά ή αστικά ζητήματα υποθέσεις της κυρίας Χάουταλα για, το πρόγραμμα, για, την έκθεση, για τη θέσπιση του προγράμματος Justice ε, υπό το άρθρο 55 του κυρίου Ράτεφ για την έκθεση περί συνεργασίας μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών ως προς την ε, καταγραφή αποδεικτικών ε, στοιχείων και τεκμηρίωση σε, αστικά ή σε εμπορικές υποθέσεις. Κυρία Χάνεμπαλ, για την έκθεση που αφορά τέσσερι αποφάσει του Συμβουλίου που επιτρέπουν σε ορισμένα κράτη-μέλη την αποδοχή τη προσχώρηση τη Δομινικανή Δημοκρατία του 100 τη Ουκρανία τη Ονδούρα στην ε, Σύμβαση τη Χάγη του 1980 για τι ε, αστικέ πτυχέ των υποθέσεων απαγωγή παιδιών, διεθνού απαγωγή παιδιών, τη κυρία Ροζιέρ για την έκθεση τη σχετική με την ε, ε, δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν της προσχωρήσεώς της στην πράξη της Γενέβης για τη Συμφωνία της Λισαβόνας σε σχέση με τις ονομασίες προελεύσεως και τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη σχετική αποφάση του Συμβουλίου του κ. Χρυσογόνου για τη γνωμοδότηση για το, ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς, της κ. Μπερζοχόν για την γνωμοδότηση σε σχέση με τη διαδικασία επαλήθευσης που σχετίζεται με τις παραβιάσεις τη νομοθεσία των κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εν τέλει του υποφαινομένου για την γνωμοδότηση τη σχετική με την ε, διακοπή της εποχιακής αλλαγής ώρας και την της απαλλαγής, σχετική με την απαλλαγή του 2017 Γενικός Προπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής δικαστήριο. Επιπλέον, οι συντονιστέ αποφάσισαν την ε, κατάρτιση γνωμοδότηση με μορφή επιστολής για την Πέτη, ε, για μια αναφορά ε, την υπαριθμό 186 του 2018, την διακοπή της προφορικής ερώτησης, τη δικασία της προφορικής ερώτησης για την οδηγία για την ασφάλεια οχημάτων με κινητήρα, ε, να ζητήσει από την νομική υπηρεσία γνωμοδότηση, γνωμάτευση μάλλον σχετικά με την ε, τροποποίηση νομική βάση της ε, πρότασης Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους καταγγέλλοντε υπαλλήλου, να αποστείλει επιστολή ο πρόεδρο σε σχέση με την πρόταση οδηγία για τη μείωση των συνεπειών και του αντικτύπου ορισμένων προϊόντων πλαστικών στο περιβάλλον, γνωμοδότηση για την ΕΝΒΗ, και να αναθέσει τον πρόεδρο να συνυπογράψει μας με τον πρόεδρο τη ΙΜΚΟ την επιστολή που αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο και που απευθύνεται στο Αυστριακή Προεδρία. Αυτό είναι το σημείο 2. Το σημείο 3 έχει να... Ε, θα έρθει αργότερα και πάμε στο σημείο 4, εξέταση σχεδίου νόμου συστάσεως για την ε, ηλεκτρονική ανάρτηση και δημοσίευση της ε, επίσημης εφημερίδας των Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητή ο υποφαινόμενο και έχω τι εξή παρατηρήσει εν ώψη της ψηφοφορία που θα ακολουθήσει αργότερα σήμερα. Έχουμε να κάνουμε με ένα, μια υπόθεση που απλώ ενημερώνει, επικαιροποιεί τον κανονισμό του 2013 για την ηλεκτρονική δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος προβλέπει και εξασφαλίζει ε, ότι η ηλεκτρονική εκδοχή της επίσημης εφημερίδας είναι επίσημη, αυθεντική, έγκυρη και ενήμερη και πλήρης έκδοση και έτσι φέρει ένομες συνέπειες. Ενώ το Κοινοβούλιο είχε χορηγήσει τη συνένεσή του για την υιοθέτηση του κανονισμού αυτού του 2013 με βάση σύσταση της Επιτροπής μας, η συζήτηση είχε εστιαστεί όχι στην ουσία της πρότασης αλλά στην νομική της βάση, που ήταν η ρήτρα ευελιξίας του άρθρου 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρήση, η επίκληση της ε, ρήτρας ευελιξίας είναι δυσκίνητη, πιθανόν και χρονοβόρα και οπωσδήποτε προβλέπεται για να χρησιμοποιείται σπάνια και κατεξαίρεση. Επιπλέον με την επίκληση τη Λίτρας αυτή στο Κοινοβούλιο μπορεί να πει μόνο ναι ή όχι, χωρίς να είναι δυνατόν να εμπλακεί στην ε, επεξεργασία του τελικού κειμένου. Επιπλέον, συνταγματικές προποθέσει ορισμένων κρατών μελών ε, επιβάλλουν και μακροχρόνιες διαδικασίες εξέτασης από τα Εθνικά Κοινοβούλια πριν την εκκίνηση ή την ε, θέση λειτουργία της ρήτρας της ευελιξίας. Η ισχύουσα τροποποιητική πρόταση έχει να κάνει με τέσσερις αιτιολογικές αναφορές και δύο σύντομα άρθρα εν ώψη των τεχνολογικών και ρυθμιστικών εξελίξεων στο ΧΕΒΙΔΕ στην επικαιροποίηση της εδικασίας του κανονισμού του 2013 για την ε, ε, πιστοποίηση της ε, γνησιότητας της επίσημης εφημερίδας μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία τώρα είναι δυνατή και με μια ηλεκτρονική σφραγίδα και έτσι επιταχύνεται η διαδικασία δημοσίευση τη επίσημη εφημερίδα. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροποποίηση αυτή είχε διατυπωθεί τον Φεβρουάριο του 2017. Η ε, Γιούρι την εξέτασε στη μορφή του κειμένου και επαλήθευσε την νομική βάση τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας το έργο της τον Σεπτέμβριο του 2017. Ωστόσο, το επίσημο αίτημα για συνένεση από πλευρά του Συμβουλίου διατυπώθηκε μόλις τον προηγούμενο μήνα. Ένα χρόνο δηλαδή, αφού του είχε κληθεί η Γιούρι να ε, διατυπώσει σύσταση για αυτή την ε, απλή επικαιροποίηση προς την Ολομέλεια στη νομοδότηση για την νομική βάση που διεκπώσαμε το 2017 και επιπλέον των, των διαδικαστικών προβλημάτων που σας περιέγραψα, είχαμε τονίσει και ε, ότι οι πιθανές τεχνολογικές εξελίξεις στη ρομποτική και την αυτοματοποίηση μπορούν να οδηγήσουν στην ε, υιοθέτηση νέων ε, πρόνοιων και διατάξεων για τη δημοσιοποίηση της επίσημης εφημερίδης και τις δραστηριότητες του, της υπηρεσίας δημοσιεύσεων που μπορεί να οδηγήσουν και σε ουσιώδεις θεμελιώδεις επιλογές ε, στην πολιτική και γι' αυτό με την ομόφωνη ε, σύστασή μας με ομόφωνη σύσταση της Επιτροπής μας απέστειλα επιστολή, ζήτησα από τον πρόεδρο Παταγιάννη, να γράψει προς το Συμβούλιο με επιστολή, δηλαδή να ζητήσει προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικέ αναθεωρήσει των συνθήκων να περιλαμβάνουν και την προσθήκη μια ρητή νομική βάση που θα εξασφαλίζει μια, ε, τη χρήση της τακτικής της ε, κοινή νομοθετικής διαδικασίας όπως ε, συνέβη άλλωστε από πάλι επιστολή λοιπόν και έτσι για το εν λόγω θέμα του Συμβούλου, έχει τυπικά ζητήσει την συνένεση με επιστολή του Κοινοβουλίου του, ε, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2018 το σχέδιο κανονισμού προβαίνει σε ίσονες αλλαγές στην πρόταση και δεν αλλάζει την ουσία της, επομένως θα επιτρέπεται η χρήση μιας ηλεκτρονικής φραγίδας για την ε, πιστοποίηση γνησιότητα τη επίσημη εφημερίδα. πρότασή μου θα ήταν προ τη Γιούρη να συσταθεί ε, στην Ολομέλεια η χορήγηση συνένεση στο σχέδιο κανονισμού. Η γνωμοδότησή μα για την νομική βάση περιλαμβάνει και τι συστάσει για την επικαιροποίηση των συνθήκων, περιλαμβάνεται στο παράρτημα που έχει προσαρτηθεί στην, ε, στο σχέδιο σύσταση. Ε, Δεδομένου και τη απλής του απλού χαρακτήρα της προτινόμενης ε, τροποποίησης της συνθήκη ε, και προκειμένου να τεθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε εφαρμογή θα πρότεινα να μην προσδιοριστεί ε, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών, να προχωρήσουμε σήμερα ακόμα το πρωί σε ψηφοφορία και να εξασφαλιστεί έτσι η δυνατότητα για έγκριση από την Ολομέλεια στη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου. Παρακαλώ τους συναδέλφους τώρα να μας κάνουν τα σχόλιά τους. Ευχαριστώ. Κανείς από ό,τι βλέπω. Η Επιτροπή θέλει το λόγο. Όχι. Έτσι λοιπόν προβλέπουμε πώς θα γίνει η ψηφοφορία για το θέμα αυτό στο, υπό το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη σήμερα το πρωί. Και συνεχίζω. Σημείο 5. Ανταλλαγή απόψεων για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα ιατρικά προϊόντα και το λόγο έχει ο κύριος Λούις Δεγράντες Πασκουάλης, ηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω να μας ακούνε με προσοχή και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η πρόταση της Κομισιόν αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και από ό,τι φάνεται είναι πολύ σωστό το και στις ρυθμίσεις. Εγώ δεν έχω καμία φιβολία για την ευκαιρία για την πρόταση, αλλά συνειδητοποιώ τις δυσκολίες που έχουμε, τις χρονικές. Εγώ άρχισα να εργάζομαι απευθείας ως συγητής ε, και φυσικά Άρχισα τις συζητήσεις με τους σκιώδεις συζητητές ε, και ελπίζω να ακούσω σύντομα τις απόψεις τους. Θέλω να υπενθυμίσω πόσο σημαντικό είναι το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασία για τη φαρμακοβιομηχανία τη Ευρώπη. Είναι μια απαραίτητη αντιστάθμιση σε όλη την ερευνητική δουλειά που γίνεται για πολλά χρόνια. Και θέλω να ξεκινήσω από εδώ, γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνία είναι το DNA τη βιομηχανία και θα πρέπει η Ευρώπη να συνεχίσει να είναι υπεύθυνη και να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα σε αυτή την καινοτομία που έχει βελτιώσει ριζικά την υγεία των ανθρώπων σε αυτόν τον αιώνα και στον προηγούμενο. Η καινοτομία σημαίνει επένδυση και ως τέτοια πρέπει να προωθηθεί και να προστατευτεί. Λαχθέντο αυτού και δίνοντα την ίδια έμφαση, υποδέχομαι θετικά την πρόταση κανονισμού σε σχέση με το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασία για τα φάρμακα, το SPC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ε, δέσμευση από την πλευρά μου να εγκριθεί στη θητή αυτή. Βέβαια γνωρίζουμε τις δυσκολίες που ενέχονται. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια συγκεκριμένη και ισορροπημένη πρόταση, όπως λέει και η Κομισιόν, στην αιτιολογική της σκέψη θέλει να καταπολεμήσει κάποιες ε, συνέπειες που προέρχονται από το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας ε, δυνάμει των αλλαγών που έζησε η φαρμακοβιομηχανία τα τελευταία 30 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντοτε κέντρο έρευνα και ανάπτυξη παραγωγή ε, του φαρμακευτικού τομέα. Εδώ αρχίσαμε το 2006 να παράγουμε βιομοειδή, δηλαδή πολύ νωρίτερα από αλλού και αυτό μετέτρεψε την Ευρώπη σε παγκόσμιο ηγέτη στην αγορά Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να υποσκάψουμε την ευρωπαϊκή ε, ανταγωνιστικότητα και να αφήσουμε σε μειονεκτική θέση τον κλάδο των γενοσύμων. Η Ευρώπη ζει σε ένα ανταγωνιστικό και παγκοσμιωμένο κόσμο, κυρίως σε αυτή την αγορά και δεν πρέπει να κόψουμε τα πόδια στις ίδιες τις επιχειρήσεις μας με στοιχεία που αφαιρούν τα κίνητρα και να χάσουμε τον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο. Εγώ θέλω να δώσω μια επικοδομητική εστίαση που να προσφέρει ασφάλεια δικαίου και εξισορρόπηση των νόμιμων συμφερόντων. Θα έχουμε μέτρα προστασίας και διασφάλισης ε, προκειμένου να καταπολεπηθούν οι, άμεσ, οι έμεσες ε, συνέπειες ε, προστατεύοντας παράλληλα την πνευματική ιδιοκτησία. Θέλουμε να έχουμε σαφήνεια και ασφάλεια και σε να δούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να ζημιωθούν οι επενδύσεις στην καινοτομία. Θέλουμε να εγγυηθούμε ότι τα εγγυώματα ε, των ε, ε, ιδιοκτών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα ζημιωθούν. Ο ρόλος των γενοσύμων φαρμάκων επίσης είναι θεμελιώδης στην εξίσωση αυτή, γιατί προσφέρουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός φάρμακα υψηλής ποιότητας με αυτόν τον τρόπο. Ε, σίγουρα έχουμε μεγαλύτερη ε, πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα αυτά και σίγουρα η εμφάνιση των γενοσύμων σήμαινε ότι οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι, πιο ευαίσθητοι, έχουν καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα. Όμως δεν θέλω να αναφέρω εδώ το θέμα της πρόσβασης στα φάρμακα, γιατί δεν συζητούμε αυτού. ούτε είναι ο σκοπός της πρότασης. Το σημαντικό είναι ότι θα δημιουργούν 20-25.000 θέσει εργασία στην ε, Ευρώπη μέχρι το 2025 και θα αυξηθούν οι καθαρές πωλήσει ε, μεταξύ 3,7 και 5,9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2025. Θα έχουμε μεγαλύτερη είσοδο των βιομοιδών και των γενοσύμων ε, στην αγορά μετά τη λήξη του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας. Επομένως, εγώ θα συνοδεύσω αυτή την πρόσταση με σημαντικές ασφαλιστικές δικλίδες ε, για να μην παρεκκλίνει σε ορισμένα σημεία, βελτιώνοντας το κείμενο της Κομισιόν, όπως παραδείγματος χάρη με κάποιες ερωτήσεις που εγώ θέλω να θέσω στην Κομισιόν, πριν να καταθέσω τις ε, τροπολογίες μου στο χρόνο που μου αναλογεί. Θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν, δεν είναι πιο λογικό μέσω στις εξάντια απαιτήσει κοινοποίηση η Παρασκευή αυτή να γίνεται από ανεξάρτητους δημόσιου φορεί καθώ και από κατόχους των δικαιωμάτων διπλωμάτων τη τεχνία και να δημοσιεύονται όχι μόνο όλα τα μέρη, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν από ανταγωνιστέ εκτός Ευρώπης για δικό τους κέρδος. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να θέσω στην Κομισιόν αρκεί ο χρόνος, 28 ε, μέρες ε, δηλαδή που δίνονται πριν ε, ως προθεσμία από την έναρξη της παραγωγής. Και τέλος, η ερώτησή μου στην Κομισιόν είναι μπορούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό ε, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την πρόταση ε, εκ των προτέρων χωρίς να ζημιώσουμε τα κεκτημένα δικαιώματα. Εδώ θέλουμε να αποφύγουμε κάποιες αρνητικές συνέπειες όπως ε, λαμβάνουν χώρα σήμερα. Είναι ερωτήσεις που ελπίζω να μπορέσει να μας απαντήσει η Κομισιόν και να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και σε σχέση με αυτά που έχω σκεφτεί, ε, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει την πρόταση τη Κομισιόν, να βελτιωθεί η πρόταση τη Κομισιόν. Σίγουρα θα ακούσω και του πιο συζητητέ και τα επιχειρήματά του. Θέλω να κάνω μια τελευταία έκκληση ότι αυτό αποτελεί μια ευκαιρία και αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να δράσουμε εγκαίρως, οι ανταγωνιστές της Ευρώπης μπορούν να ε, καλύψουν ε, το δικό μας χώρο και μπορούν να ζημιώσουν όχι μόνο το χώρο των γενοσύμων αλλά και το χώρο της καινοτομία. και τελικά ο ασθενής θα είναι αυτός που θα πληγεί. Όμως ε, είναι κάτι πολύ απλό αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κατάσταση καταξαίρεση έτσι ώστε τη μέρα που θα πολλούνται τα γενώσιμα να μην μας πάρουν τη θέση οι ανταγωνιστές της Ευρώπης και να μπορούμε να ανταγωνιστούμε συνοχίζοντας να είμαστε σε πρώτη ηγετική θέση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βόλκεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, παρουσίασή του και τα πολύ θετικά του λόγια για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ μαζί του. Θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ένα καλό πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και αρκετό καιρό έχει ζητήσει ε, να παρέχονται κίνητρα για την πρόσβαση στα φάρμακα. Από το 2016 ξεκινήσαμε τις εργασίες μας και πέρυσι είχαμε την ε, έκθεση για την καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα. Εμείς ως ε, νομοθέτης, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να ε, γίνεται έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων. Βλέπουμε ορισμένα παραδείγματα όπως τα της Δανίας για παράδειγμα που είναι πολύ ισχυρή ε, δύναμη στον χώρο των γενώσιμων φαρμάκων και είναι πρωτοπόρος στην ε, φαρμακευτική καινοτομία. Γι' αυτό θα ήθελα να στηρίξω απόλυτα τον εισηγητή και τις σκέψεις του ότι η νομοθεσία θα μας οδηγήσει σε κάτι πολύ θετικό. Ε, φυσικά οι αλλαγές γίνονται ταχύτατα, εξελίσσονται τα πράγματα πολύ γρήγορα και ε, είτε τα γενώσιμα φάρμακα είτε, είτε τα βιοομοειδή ε, είναι κατηγορίες που πρέπει να παρακολουθούμε συνέχεια και να τροποποιούμε την νομοθεσία καταλήλως. Χρειάζεται να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Με τον κανονισμό αυτό θα, δημιουργηθεί, θα δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις εταιρείε με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις εξαναγωγές τους σε χώρες που δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις για τα, ε, τις κατηγορίες αυτές φαρμάκων ούτε και, και επίσης θα προστατευτεί η πνευματική ιδιοκτησία. Τα SPC δεν θα, ε, και δεν θα επηρεάζονται από την ε, θέση ισχύ του κανονισμού. Η διάρκεια ισχύς προβλέπεται στα πέντε χρόνια και η εισαγωγή επίσης γενώσιμων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική ε, διότι μπορεί να μειώσει τις ε, τιμές των φαρμάκων και να ε, έχει αυτό θετικά αποτελέσματα για τον προϋπολογισμό των κρατών. Τώρα, η είσοδος στην... σε ό,τι αφορά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ πως, πως δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν εξαιρέσεις μόνο για τις εισαγωγές αλλά και για την αποθήκευση, stockpiling. Νομίζω πως με τις προσθήκες και τις οπλίσεις αυτές ε, η πρόταση αυτή θα αξιοποιήσει όλες τις ε, δυνατότητες που έχει έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε τα φάρμακα αυτά να μην ε, παράγονται σε ξένες χώρες και να καθιερωθεί η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη ως ε, πρωτοπόρος και να μην υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ. η Ιαπωνία. Θα καταθέσω ορισμένες τροπολογίες οι οποίες ελπίζω να επηρεάσουν θετικά ε, την έκθεση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα προτείνω ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες, ε, Σύμφωνα με την οδηγία για τα φαρμακευτικά σκευάσματα, επίσης ε, τροπολογίες σχετικά με την υποχρέωση κοινοποίηση. Η προθεσμία των 28 ημερών θεωρώ πως ε, είναι αρκετή. Θα μπορούσαν να είναι αρκετές και 14 μέρες ε, για να κοινοποιούνται οι αρμόδιες αρχές και με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να προστατευτούν και τα εμπορικά συμφέροντα. Επίσης, ε, θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες για την αποθήκευση φαρμακευτικών σκευασμάτων. Τώρα, η αποθήκη, υπάρχει το επιχείρημα πως δεν, ε, μπορεί, δεν μπορούν να αποθηκεύονται φάρμακα διότι αυτό αντιτίθεται σε ορισμένε εμπορικέ πρακτικές. Δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτήν την άποψη. θεωρώ πως ε, πολιτικά θα είναι ζήτημα που θα διχάσει. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές και να ευχαριστήσω όλους για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζλωτόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε. Κάποια σχόλια για την πρόταση. Η φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική και να ανταγωνίζεται με ίσους όρους ε, σε σχέση με τις άλλες χώρες όσον αφορά τα γενώσιμα φάρμακα. Η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία έχει υψηλά πρότυπα ασφάλειας και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πρότυπα αυτά προς όφελος των καταναλωτών και των καταναλωτών ε, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και αλλού. Μέχρι το 2020 θα υπάρχουν φάρμακα χωρίς προστασία αξίας 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κανονισμός λοιπόν οφείλει να αλλάξει έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας στην ε, διεθνή αγορά. Φυσικά όμως χρειάζονται και νομικές ασφαλιστικές δικλίδες που θα προστατεύουν από κατάχρηση. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται επίσης όμως να παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής των προϊόντων αυτών για εξαγωγές ο ανταγωνισμός από την Κίνα και τη Ρωσία είναι πολύ μεγάλος και η πρόταση αυτή θα μας δώσει μια μεγάλη ευκαιρία να προσελκύσουμε επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. που θα βοηθήσει πολύ και τον τομέα των καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων, θα συνεισφέρει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και μεταφοράς γνώσης. Η ομάδα μας είναι υπέρ της πρότασης της Επιτροπής. Έχουμε όμως κάποιες επιφυλάξεις ως προς το ποια από αυτά τα SPC, αυτά τα σκευάσματα, θα ε, συμπεριλαμβάνονται και ποια θα είναι η χρονική τους διάρκεια. Αυτό νομίζω θα καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία της πρότασης. Θα καταθέσουμε λοιπόν ε, τροπολογίες και ελπίζουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως κάθε φορά που εξετάζουμε τέτοια ζητήματα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι όταν τροποποιούμε κανονισμούς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θέσουμε σε κίνδυνο δικαιώματα για ε, την προστασία των ε, επιχειρήσεων των εσκευασμάτων αυτών, τα οποία είναι τεχνολογίας εχμής, είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Ο κανονισμός αυτός θα βοηθήσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο σταθερό πλαίσιο για την φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη και θα δημιουργήσει ίσως όρους ανταγωνισμού ε, σε σχέση με τις άλλες εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Εταιρείε που δραστηριοποιούνται εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα έχουν την δυνατότητα να διαθέτουν τα γενώσιμα φάρμακά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νωρίτερα από την ημερομηνία που θα τα διαθέτουν οι εταιρείε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Χρειάζεται προστασία και ο κανονισμό θα βοηθήσει σε αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι η ποιότητα των ε, φαρμακευτικών προϊόντων είναι πολύ σημαντική για τους καταναλωτές. Υπάρχουν και τα πλαστά φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δυστυχώς κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά και τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από την Κίνα. Όχι και διατίθενται όχι μόνο μέσω του διαδικτύου, αλλά και μέσω ύποπτων φαρμακείων. Δυσκολεύομαι λοιπόν να κατανοήσω τα κίνητρα πίσω από αυτές τις δραστηριότητες, διότι είναι καταστρεπτικές οι συνέπειες που έχουν για την υγεία. Επίσης, χρειάζεται προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό εξάλλου είναι καθήκον μας. Τα δύο αυτά βασικά θέματα με τα οποία καταπιάνεται ο κανονισμός πρέπει να έχουν και, τις ε, κατάλληλες, ε, και το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα. Και πρέπει ο κανονισμός να συμπεριλαμβάνει και φάρμακα τα οποία δεν έχουν παρασκευαστεί, δεν έχουν συνδεθεί ακόμα, διότι η τεχνολογία εξελίσσεται. Μετά, έπειτα από την λήξη της ε, περίοδου των 5 ετών, οι εταιρείε από τρίτες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω πως αυτό θα είναι ε, αμοιβαία επωφελές και για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ε, εταιρείε από τρίτες χώρες. Οι ευρωπαϊκές εταιρείε δαπανούν τεράστια ποσά για έρευνα και ανάπτυξη και φυσικά είναι υπέρ μιας ε, πρόσθετης ε, περίοδου προστασίας 5 ετών και ασφαλιστικών δικλείδων. Οι ευρωπαϊκές φαρμακευτικές ε, επιχειρήσεις παράγουν προϊόντα άριστης ποιότητας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να τις προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει να αντιδράσει. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την ευκαιρία που μας ε, δίνετε να τη δράσουμε σήμερα το πρωί. Μπορώ να διαβεβαιώσω τον εισηγητή για δύο πράγματα. Καταρχήν, ακούσαμε πολύ προσεκτικά όλα όσα υπόθηκαν σήμερα το πρωί και είμαστε ικανοποιημένοι που ακούμε ότι υπάρχει θετικό πνεύμα απέναντι σε αυτή την πρόταση. Δεύτερον, ναι, βεβαίως είμαστε στην πλήρη διάθεση της Επιτροπής σας προκειμένου να βρούμε λύση για να παρασχεθεί η τεχνική βοήθεια που χρειάζεται. Ευχαριστώ να το κάνω αυτό. Όπως υπογράμμισε ο εισηγητής, η πρόταση αυτή όντω προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες, είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό, για τις ευρωπαϊκές εταιρείε, προκειμένου να δράξουν τα ωφέλη σε αγορέ που μεγενθύνονται ταχύτατα. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την πρόταση και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και φυσικά θα προσφέρουμε την πλήρη μα βοήθεια. Καθώ χρειαζόμαστε αυτή την πρόταση τώρα και καθώ πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, όπω τόνισε και ο συγητής, ο στόχο μας ήταν να καταθέσουμε μια στοχευμένη πρόταση και περιορισμένη και, και να έχουμε και μια ισορροπημένη προσέγγιση, να μην κάνουμε παραπάνω από όσα χρειάζονται προκειμένου να βοηθήσουμε τις εταιρείε βιομοιδών και γενοσύμων με βάση την Ευρώπη να αδράξουν τα ωφέλη των ε, παγκόσμιων αγορών που μεγενθύνονται γρήγορα. Αυτό ήταν ο στόχο τη Επιτροπή και χαίρομαι που, της πρότασης, συγγνώμη, και χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχει υποστήριξη για την πρόταση αυτή. Τώρα, να έρθω στι συγκεκριμένε ερωτήσει που τέθηκαν. Αν κατάλαβα καλά την πρώτη ερώτηση του συγητή το θέμα της απέτησης κοινοποίηση. Και η ερώτηση είναι γιατί θα πρέπει να γίνει, δίνονται οι πληροφορίες αυτές στον κάτοχο του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασία. Θα σας εξηγήσω την, την προσέγγισή μας. Η προσέγγισή μας ήταν να παρέχουμε κάποιες πληροφορίες ε, μέσω των εθνικών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνία που υποχρεούνται να δημοσιεύσουν αυτές τις πληροφορίες ε, και προσωπικά και προσεκτικά διαμορφώσαμε τις προτάσεις έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν διαβιβάζονται εμπιστικές πληροφορίες ε, άμεσα στους κατόχους ε, του SPC. Λεχθέντος αυτού, θα διερευνήσουμε φυσικά πιθανές λύσεις στον τομέα αυτό. Όμως η ανάγκη να προστατεύσουμε τις της πληροφορίες φαίνεται να είναι πολύ σημαντική. Δεύτερον, τα στοιχεία τα χρονικά. Αν άκουσα καλά, ο εισηγητή πιστεύει ότι οι προθεσμίες που βάλλονται σε διαδικασία κοινοποίηση είναι κάπως φιλόδοξες και άκουσα ότι ο σκιώδης εισηγητή είχε διαφορετική άποψη. Και πάλι αυτό είναι ένα θέμα επί το οποίο ευχαριστώ να προσφέρουμε τεχνική βοήθεια. Θέλαμε μια προθεσμία που να είναι ρεαλιστική και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και των δύο πλευρών. Τρίτον, Τώρα, η εφαρμογή της πρότασης σε χρόνο. Πράγματι, η πρόταση της Κομισιόν σκοπεύει να διασφαλίσει ότι η απαλλαγή θα ισχύσει για συμπληρωματικά πιστοντικά προστασία που δεν έχουν χορηγηθεί ακόμα την, ε, την ημερομηνία της θέσης ισχύ του κανονισμού. Με μια πολύ περιορισμένη με ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Γιατί επιλέξαμε αυτή τη λύση. Υπάρχουν πολλέ λύσει δυνατέ. Εμεί επιλέξαμε τη λύση αυτή βάσει μια αξιολόγηση αναλογικότητα. Αφενό, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις μας μπορούν να υποφεληθούν το συντομότερο από τα ωφέλη της απαλλαγής, γιατί επίκειται η λέξη πολλών διπλωματών τεχνίας. Απ' την άλλη, είμαστε προσεκτικοί ότι τα προστατευόμενα δικαιώματα γίνονται σεβαστά όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν και πάλι βρήκαμε αυτή την ισορροπία και ευχαριστώ να προσφέρουμε τεχνική βοήθεια γιατί ακούσαμε εδώ στην αίθουσα ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. για το επιχείρημα σε σχέση με την εφαρμογή στον χρόνο ότι αυτό οδηγεί σε διαφοροποιημένες εφαρμογές ε, στην Ευρώπη αυτή η διαφοροποιημένη εφαρμογή είναι εγγενής στο σύστημα SPC. Εξαρτάται που θα καταθέσεις την αίτησή σου και κατόπιν εξαρτάται από το τι θα κάνει το Εθνικό Γραφείο Διπλωμάτων Τεχνίας. Έτσι λοιπόν ένας ε, βαθμός ε, διαφοροποίησης υπάρχει ήδη και σήμερα. Αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερα προβληματικό λοιπόν. Τώρα, για να αναφερθώ σε κάποιες δηλώσεις του κ. Βόλκα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία. Αν κατάλαβα καλά, θέλετε να προωθήσετε ένα σύστημα που θα ισχύει μια απαλλαγή όχι μόνο για την εξαγωγή εντός, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε εξαγωγές εντός της Ένωσης, εκεί όπου δεν υπάρχει προστασία του SPC. Εμείς θεωρούμε ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα, γιατί βλέπουμε ότι αναπτύσσονται παντού τα SPC και υπάρχει αυξανόμενη χρήση του. Έτσι λοιπόν, δεν είμαι τόσο σίγουρη ποια θα ήταν η προσθέμενη αξία. Αλλά να το διερευνήσουμε. Είμαστε πρόθυμοι. Τώρα, ο κ. Βάλκαν τόνισε την ανάγκη να διευκολυνθεί εξ αρχή είσοδο για τα γενώσιμα και τα βιομοειδή. Δηλαδή εξ αρχή είσοδος στις ευρωπαϊκές αγορές όταν ε, λύγει η προστασία SPC. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και πιστεύουμε ότι η πρότασή μα όντω θα διευκολύνει την είσοδο από την πρώτη μέρα. Και είναι πολύ απλό ο λόγο. Αν μπορεί ε, να παρασκευάσεις στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της περίοδου προστασίας SPC, τότε έχεις ικανότητες παρασκευής και είναι πιο εύκολο να εξάγεις εκτός. Από ό,τι βλέπω, τελειώνω χρόνος μου, θα είμαι πολύ γρήγορη. Δύο λόγια για την αποθήκευση. Καλό τους συζήτητες να δουν τη μελέτη αντικτύπου. Εκεί αναφέρονται πολλοί λόγοι γιατί η Κομισιόν δεν έχει συμπεριλάβει στην πρόταση την αποθήκευση, αλλά θα σταματήσω εδώ γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ και λυπούμε που σας διακόπτω. Ελπίζω να έχουν δοθεί απαντήσεις, κυρίως προς τον εισηγητή. Κύριε Πασκουάλη, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα Χαίρομαι που βλέπω ότι η στάση απέναντι σε αυτή την πρόταση θα μας επιτρέψει να βρούμε μεγάλους συμβιβασμούς. Εγώ θεώρησα ότι βρίσκω τον εαυτό μου στα λόγια όλων. Είναι πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και μπορούμε να συμπληρώσουμε και να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν, αλλά δεν υπάρχουν ε, μεγάλες διαφοροποίησεις. Ε, μας ε, ενώνει το πνεύμα βελτίωση. Βέβαια, θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα τη αποθήκευση και με την Κομισιόν, όμω είναι μια εξαιρετική στιγμή ευκαιρία που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη σχόλιά τους, ευχαριστώ και την Κομισιόν και ελπίζω να συνεργαστούμε με επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ως εκ τούτου, το σημείο 6. Εξέταση τροπολογιών για διασυνοριακές ε, μετατροπές, χωνεύσεις κτλ. Ακολουθεί η κυρία Ρέγνερ, έχει το λόγο η συγγήτρια. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Οι τροπολογίες σας τώρα έχουν από την τρίτη μεταφραστή και είναι στη διάθεσή σας στα αγγλικά. Είναι πάνω από 800, γι' αυτό το επισημαίνω μόνο οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί σε εμά. Ακολουθούν ε, η ΕΚΟΝ και η ΕΜΠΛ ένα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα στην ΕΚΛ η δουλειά γίνεται μόνο στα αγγλικά για να μπορούν γρήγορα να προχωρήσουν και με δεδομένη τη στενότητα θέλουν να, χρόνο θέλουν να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Ε, σήμερα λοιπόν έχουμε μια πρώτη συνάντηση σκιωδών την οποία περιμένω με χαρά. Όμω είχα και την ευκαιρία και θα έχω και στο μέλλον να συνεχίσω και τι διμερεί επαφέ που είναι πολύ επικοδομητικές. 19 με 20 Νοεμβρίου προβλέπεται η ψηφοφορία. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω, να πιεστώ δηλαδή χρονικά για ε, να είμαι έτοιμη με δεδομένα τα χρονικά περιθώρια και το περίπλοκο του θέματος. Αυτό μπορώ να πω προκαταβολικά για τις τροπολογίες είναι ότι από όλες τις ομάδες βλέπω το αίτημα για ένα νέο νομικό πλαίσιο, μια σαφή διαδικασία που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις την κινητικότητα μέσα στην ενιαία αγορά χωρίς να πρέπει να αλλάζουν νομική προσωπικότητα ή να εγκαταλείπουν νομική προσωπικότητα αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας και όρους ασφάλειας δικαίου. Αυτή είναι η κυρία απέτηση αυτή τη στιγμή. Και οι κύριοι παράγοντες φορείς όπως εργαζόμενοι, όπως ε, πιστωτές και όπως λοιποί φορείς πρέπει να προστατεύονται. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε το εταιρικό δίκαιο και μια εξέλιξη η οποία οδηγεί στο να μην υπάρχει μέχρι τώρα προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αναμετατροπή συγχώνευση κτλ. ή τουλάχιστον αυτή η προστασία να εναπόκειται μόνο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε αυτό ε, θεωρούμε ότι το λεγόμενο forum shopping, δηλαδή η αναζήτηση της πιο ευνοϊκής δικαιοδοσίας έχει οδηγήσει σε πολλά προβλήματα και εντάσεις μεταξύ των κρατών μελών και ε, εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι εντάσεις. Επομένως χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες, σαφείς διαδικασίες και υψηλό επίπεδο προστασίας των εμπλεκομένων πλευρών, κυρίως των εργαζομένων που πλήττονται από αυτές τις μετατροπές, συγχωνεύσεις κτλ. Τώρα, τροπολογίες θα είμαι πολύ ε, λακωνική γιατί ξέρω ότι έχουμε λίγο χρόνο μέχρι ότου ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες μας αλλά είναι και πολλές και περίπλοκες οι τροπολογίες ε, με σημασία ορισμένες ε, κέρια. Οι τροπολογίες μας λοιπόν των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την προστασία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων αυτών έχουν κατατεθεί ε, περιλαμβάνουν όρους ενημέρωσης διαβούλευσης αλλά και συναπόφασης με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο, προσαρμογή δηλαδή του κεκτημένου και αντίστοιχη προσαρμογή των ευρωπαϊκών καθεστώτων που θα πρέπει να εξασφαλίσουν έτσι δικαίωμα στην απόφαση του εργαζομένου προς μέσα σε επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα προβλέπεται η διευκρίνηση πως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμετέχουν σε διοικητικά όργανα ε, για την λήψη των αποφάσεων. Συνεχίζω και αναφέρω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επιχειρήσεων ή το Σωματείο των Εργαζομένων, μέσα από το οποίο εκπροσωπούνται αυτοί, πρέπει να έχει και τους απαραίτητους πόρους στη διάθεσή του για να αναλύει την έκθεση περί συγχώνευσης και ούτω καθεξής και ταυτόχρονα οι διαβουλεύσεις ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουν το δικαίωμα για τον εργαζόμενο, τους εργαζομένους, να λάβουν μία απάντηση στα ερωτήματά τους πριν να ληφθεί η απόφαση. Γιατί βλέπουμε ότι πολύ συχνά μπορεί να εμφανίζεται μια απάντηση, αλλά να έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, δηλαδή έχουν εγκριθεί και αποφασιστεί τα πάντα. Επομένως θέλουμε μια έγκαιρη απάντηση. Για τις λοιπές τροπολογίες τώρα. ο ορισμός της ε, εταιρείας γραμματοκιβωτίου ή των λεγόμενων τεχνητών διευθετήσεων πρέπει να βελτιωθεί. Απαιτούμε μέσω της, ε, του σχεδίου εκθέσεις μια ουσιαστική δραστηριότητα της επιχείρησης στο κράτο μέλος στο οποίο θα καταχωριστεί αυτή. Δεν θέλουμε δηλαδή να υπάρχουν μόνο εικονικές έδρες σε χώρες ε, του εξωτερικού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και οι εικονικές λειτουργίες όπως τις αναφέρουμε σημαίνουν ότι θέλουμε να έχουμε πραγματικούς φορείς της οικονομικής δραστηριότητας μέσα στα κράτη-μέλη και για αυτούς να προβλέπεται η κινητικότητα και η δυνατότητα διαφύλαξης των δικαιωμάτων τους. Πολλές ομάδες επίσης έχουν καταθέσει τροπολογίες ζητώντας η, έδρα, καταστατική έδρα και η διοικητική έδρα να είναι στην ίδια χώρα. Την υποστηρίζω την πρόταση αυτή και θα ήθελα επίσης από τους συντάκτες της σχετικής τροπολογίας ε, πιο πολλές λεπτομέρειες για, τα, ε, για τη λογική του, της τροπολογίας και το στόχο της. Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε φαντάζομαι στις ε, συναντήσεις των σκιωδών. Για το άρθρο 86F έχουμε τροπολογία από πολλές ομάδες ε, που έχουν να κάνουν με συμπλήρωση της διατύπωσης. Θεωρώ ότι βελτιώνουν το κείμενο και τις υποστηρίζω. Έχουμε επίσης τροπολογίες που στοχεύουν στην απλούστευση της διαδικασίας της έκθεσης περί συγχωνεύσεως ε, κτλ. Ε, δεν θα επεκταθώ, είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε ούτως ή άλλως με τους και στη συνάντηση που θα γίνει σήμερα ε, και αναλόγω, βέβαια θα διευκρινίσουμε και κάποια ζητήματα και ενδεχομένω θα τα ομαδοποιήσουμε. Θα ήθελα να καταλάβω περισσότερο τι συνέπειες, τι κόστο ε, τι απόδοση μπορεί να έχει μια τέτοια πρόταση και επίση θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπολογίε αυτέ που αναφέρονται σε ανεξάρτητους πραγματογνώμονε όπου έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Βεβαίω υπάρχει μια σειρά από δυνατότητε που προτείνουν οι τροπολογίε για ανεξάρτητου πραγματογνώμονε. δύο λένε άλλοι, κάποιοι άλλοι λένε όχι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις δημόσιες αρχές, ε, μπορούν να ε, κάνουν μια ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση και αν χρειάζεται να προσταθούν σε αυτές και οι ανεξάρτητοι πραγματογνωμόνες. Αλλά ε, με, όλο το, με όλη την κατανόηση που έχω για την λογική αυτών τροπολογιών δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι υπάρχει και η ανάγκη για την ασφάλεια δικαίου στο σύστημα που θα ισχύει. Αυτό λοιπόν πρέπει να διευκρινίσουμε και ενδεχομένως ε, τα ζητήματα αυτά που ίσως να μπορέσουν να ξεκαθαριστούν ε, τώρα μπορούμε να τα δούμε βέβαια στην, ε, στη συναντήση των σκιωδών. Ευχαριστώ Τυρό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και πολύ σύντομα για να ευχαριστήσω καταρχάς την Εύλην για τη δουλειά που έχει κάνει στην ε, στο σχέδιο αυτό εκθέσεω, για να εξηγήσω λίγο τι τροπολογίε μα. Θα, θα πω καταρχά ότι συμφωνούμε επί τη αρχής, επί της αρχής. Στη διατύπωση ίσως να υπάρξει κάποια διευκρίνηση, κάποια αλλαγή. Λέτε εσεί ότι πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο οι εργαζόμενοι και δει τα σωματεία τους ε, στις ε, υποθέσει αυτέ, συγχώνευση κτλ. Ε, εμείς αυτό που θα θέλαμε θα ήταν να ενισχύσουμε την αρχή του ανελκυστήρα, δηλαδή οι μικρές επιχειρήσεις να μην εκτίθενται στην ίδια νομοθεσία, στις ίδιες διατυπώσεις δηλαδή με αυτές που ισχύουν για τις μεγαλύτερες, έτσι ώστε να έχουμε και μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος. Αυτό επίσης το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το ζήτημα της γνήσιας έδρας, της πραγματικής έδρας, για να μην έχουμε απάτες, για να μην έχουμε κάτα καταστρατήγηση του δικαίου και πλασματικές έδρες ή μετατοπίσεις, προκειμένου φερειπίν κάποιο να αποφύγει τη φορολογία ή τις ε, ε, εργοδοτικές εισφορές. Ε, αυτά νομίζω μπορούν να διευκρινιστούν και επίσης θα θέλαμε όλες αυτές οι εξαγορές, ε, συγχωνεύσεις, μετατροπές λοιπά, να καλυφθούν να καλυφθεί εξ ολοκλήρου χωρίς να υπάρχουν γκρίζες ζώνες ή ασάφειες για το ποιες είναι οι δραστηριότητες συγχώνευσης και το καθεξής που υπάγονται στο νομοθέτημα. Αυτό. σα έχουμε δώσει τροπολογίε. περιμένουμε τη συζήτηση και βεβαίως είμαστε υπέρ τη απλοποίηση των διαδικασιών. Κύριος Δεγράντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κινηθούμε γρήγορα και να μην καθυστερήσουμε στην πρώτη αξιολόγηση των ε, τροπολογιών. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε χρόνο. Επομένως, ε, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε τις απόψεις μας ε, σε σχέση με τις τροπολογίες τόσο της εισηγήτριας όπως και των υπόλοιπων σκιωδών. Απλώς θα πω κάποια γενικά σχόλια. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρέγκνερ, την εισηγήτρια, για την ευγενική της τάση, είναι μέρος της προσωπικότητάς της. Εμείς ε, λεπτομερώς στη συνάντηση των σκιωδών θα ανταλλάξουμε απόψεις. Πάντως ευχαριστώ και το έργο των υπολείπων, συγητών. Μπόρεσα να διαβάσω τις εκθέσεις και απλώς θέλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Εγώ πιστεύω ότι ο στόχος ε, δεν θα πρέπει να είναι να αυξήσουμε το διοικητικό άχθος των εταιριών, γιατί αυτό θα χειροτερεύσει την νομοθεσία και μάλιστα ε, δεν ε, θα βοηθήσει στην ε, αύξηση της αντιγωνιστικότητας. Πρέπει να προωθήσουμε την επικουρικότητα, το να διευρύνουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων πέρα από αυτό που προβλέπεται στην αρχή πρώτης Κομισιόν αποτελεί λάθος. Υπάρχει ο μηχανισμός διαβούλευσης, ενημέρωσης και συμμετοχής των εργαζομένων Το να αυξήσουμε απλώς αυτό θα αποτελούσε διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις. Αυτό που έχουμε βέβαια ε, στην έκθεση της εισηγήτριας είναι λογικό. Γιατί οι μετατροπές συγχωνεύσεις και διασπάσεις σε διασυνοριακό επίπεδο μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σίγουρα θα χρειαστούν ασφαλιστικές δικλείδες ε, για ε, κάποιες έκτακτες περιπτώσεις. Σε αυτό θα συμφωνούσα. Όμως ε, δεν θα ήθελα τώρα να αλλοιώσουμε το ότι υπάρχει ήδη σε άλλες οδηγίες και να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία χωρίς να είναι απαραίτητο. Ξέρετε ποια είναι η στάση μου κύριε Ρέγνερ. Είμαι υπέρ στο να βρούμε μια συνένεση σε όλες αυτές ε, τις ε, θέσεις και νομίζω ότι με καλή πίστη θα συνεργαστούμε για να βρούμε τους απαραίτητους συμβιβασμούς, τις απαραίτητες συμφωνίες. Φυσικά θα ακούσω και τις πρωτοβουλίες των επόμενων σκιωδών και ίσως να μπορέσουμε να βρούμε μια ικανοποιητική λύση που να εγγυάται οι νέε κινήσει των επιχειρήσεων, οι νέε καταστάσει που μπορούν να συμβούν σε παγκοσμιοποιημένο κόσμο να είναι καλέ για την επιχείρηση και για τη δημιουργία θέσεων εργασία και ε, ταυτόχρονα δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους. Επίσης, ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα αποφεύγονται και οι απάτες θα πρέπει βέβαια να είμαστε καλόπιστοι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να προσφέρουμε ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι πολλά πράγματα θα πρέπει να τα αφήσουμε και στα κράτη-μέλη, να διαφυλάξουμε την επικουρικότητα. Να μην είναι εξαντλητικό ο ρόλο τη Ευρώπη και να μπαίνει σε χωράφια που δεν τις αρμόζουν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαρίνο Επίντου. Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω μια διαμαρτυρία. Γιατί δεν έχω εδώ διερμηνία. Δεν είναι εδώ η ομάδα της διερμηνίας. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα μου, ούτε μπορώ να ακούσω τις παρεμβάσεις των συναδέλφων στη δική μου γλώσσα, στα πορτογαλικά. Είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη σήμερα εδώ. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Χρειάζεται περισσότερο σεβασμό για τους βουλευτές. I fully agree with you. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν μας ενημέρωσαν πως δεν θα υπάρχει διερμηνία στην πορτογαλική γλώσσα. Γι' αυτό λοιπόν ε, είμαστε μαζί σας, να το ξέρετε. Δεν μπορώ να μιλήσω πορτογαλικά γιατί δεν υπάρχει διερμηνία. Ε, on vient Μόλις μας είπαν ότι μπορείτε να μιλήσετε. Μπορείς να μιλήσεις πορτογαλικά. Α, μπορώ να εκφραστώ, αλλά δεν μπορώ να ακούσω. Μάλιστα. Αλλά ισχύει η διαμαρτυρία, γιατί οι διερμηνείς έφυγαν. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ε, thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Εύελιν. Πολύ σωστά οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, ωστόσο πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο ε, το οποίο θα διέπεται από διαφάνεια, από σοβαρότητα, συνέπεια και θα ε, βελτιώσει την ε, ενιαία αγορά. Γι' αυτό προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της πραγματικής έδρας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την καταστατική τους έδρα σε ένα άλλο κράτος μέλος μόνο εάν μεταφέρουν και την πραγματική τους έδρα εφόσον δηλαδή μπορούν να αποδείξουν ότι ε, έχουν ουσιαστικές οικονομικές δραστηριότητες στο κράτος προορισμού και, θα, και χρησιμοποιούν ε, τις ε, δυνατότητες που έχουν για ελευθερία εγκατάστασης. Χρειάζεται λοιπόν ισχυρή και αυστηρή αρχή πραγματικής έδρας έτσι ώστε να ε, αποτραπεί η δημιουργία εταιριών βιτρίνων. Θεωρώ λοιπόν πως έτσι θα βελτιωθεί η πρόταση. Επίσης, η πρόταση για... οι προτάσεις για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τα σχετικά δικαιώματα χρειάζονται βελτιώσεις έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να επηρεάζουν τις αποφάσεις της διοίκησης. Η εταιρική κινητικότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβούλευση και επαρκή εκπροσώπηση, γι' αυτό χρειάζεται τα πρότυπα να ενισχυθούν και όχι να αποδυναμωθούν. Ο κύριος Φως και ο κύριος Ντεγκράντες Πασκουάλ από το ΕΛΚ έχουν προτείνει μια τροπολογία επανεισαγωγής συγκεκριμένων ανώτατων ορίων για τον αριθμό των εργαζομένων στην συμμετοχή στα Συμβουλία Επιχειρήσεων. Αυτό είναι σύμφωνο με τις γερμανικές πρακτικές. Ωστόσο, στη Σουηδία υπάρχουν αυστηρότατοι κανόνες για τη συμμετοχή των εργαζόμενων, ακόμα και σε εταιρείε που έχουν πάνω από 25 υπαλλήλου. Ε, αυτή η πρόταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμά. Τη θεωρούμε παράδεκτη διότι θα βλάψει ε, πολύ το σύστημα της ιδέας. Επίσης, να πω ότι η πρόταση αυτή είναι μία από τις δύο νομικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου και πρέπει να την ε, κρατήσουμε και να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, διότι πρέπει να, συνοδεύω, να συνοδεύει με την άλλη στις διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Να είστε σύντομοι όμως, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, ταχεία πρόοδο στην κατάρτιση της έκθεσης και να ευχαριστήσω και όσους κατέθεσαν τροπολογίες για αυτό το αρκετά περίπλοκο θέμα. Από τον αριθμό τους καταλαβαίνω ότι Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την πρόταση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να βρει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και την διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ε, επιχειρήσεων. Αυτό ανέφερε και η συγγήτρια εξάλλου. Πώς δηλαδή μπορούμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις, ταυτόχρονα όμως ε, διατηρώντας ασφάλεια δικαίου και οι προτάσεις ε, αυτές μας βρίσκουν σύμφωνος. Έχουμε καταφέρει να βρούμε μια σχετική ισορροπία, όμως ε, χρειάζεται διαπραγμάτευση σε πολλά σημεία. Με χαρά μας λοιπόν να συνεργαστούμε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να βρεθούν τεχνικές λύσεις. Να τονίσω επίσης ότι με την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους υφιστάμενους κανόνες για τις μετατροπές και τις ε, συγχωνεύσεις. Οι διαιρέσεις ε, θα είναι ένα νέο στοιχείο που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες οι μορφές εταιριών. Θα πρέπει επίσης να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις μετατροπών συγχωνεύσεων και διαιρέσεων για να μην μπορεί να γίνει παράκαμψη των κανόνων και να μην μένουν ανοιχτά παραθυράκια. Χρειάζεται να καλύπτονται και οι μετατροπές και οι διαιρέσεις από τη νέα πρόταση. Τώρα, η επιλογή των συγκεκριμένων λύσεων βασίστηκε στην ομολογία πριν την υποβολή της ε, πρότασης από εμά. Γι' αυτό η Κομισιόν δεν πρότεινε την αρχή της πραγματικής έδρας για κάθε περίπτωση, γιατί θεωρούμε πως αυτό δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την ομολογία. Και να πω στην συνάδελφο ότι όλα τα κράτη-μέλη τα οποία εφαρμόζουν την αρχή της πραγματικής έδρας που απαιτεί η, η εταιρεία να έχει την πραγματική της έδρα εκεί όπου δραστηριοποιείται μπορούν να την ε, διατηρήσουν ακόμα και μετά την πιθανή έγκριση της πρότασης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια για τους εργαζόμενους, εμείς επιλέξαμε ένα αναλογικό σύστημα για να ληφθούν υπόψη και οι κανόνες ε, όλων των κρατών μελών για τη συμμετοχή των εργαζομένων. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησαμε την αρχή των τεσσάρων πέμπτων. Να κλείσω λέγοντας πως ε, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Ο Νοέμβριος ε, μας ικανοποιεί πολύ διότι θεωρούμε ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με τις ε, νομοθετικές αυτές προτάσεις ως σύνολο και με τις δύο ταυτόχρονα. Αυτός είναι όντως ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί. Καλώς σας ευχαριστώ. Στα πρακτικά, όπω είπε η συγγήτρια, 19 Νοεμβρίου προβλέπεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή μα. Θέλετε πάλι το λόγο, κυρία Ρέγνερ. Ναι, ξέρω ότι έχουν έρθει όλοι έτοιμοι και περιμένουν την ε, ψηφοφορία. Απλώ ε, για να ολοκληρώσουμε ε, και μια και συζητήθηκαν διάφορε πτυχέ, θα τονίσω ότι θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, να, προχωρήσουμε, να προωθήσουμε γρήγορα και τους δύο φακέλους, αυτό το έχουμε πει. Η ταχύτητα σημαίνει βέβαια μάλλον ταυτότητα δεν σημαίνει ότι ε, κάνουμε στο πόδι της, ε, την επεξεργασία και τις ρυθμίσεις. Ξέρουμε ότι στις λεπτομέρειες κρύβεται ο σατανάς και πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς, με πολύ ακριβές, δια, διατάξεις, στην ώρα μας βέβαια να ολοκληρώσουμε, αλλά και να σεβαστούμε και να εξασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Ζήτησε επίσης το λόγο διότι θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω αυτό που είπε ο κύριος Μαρίνιο Τιπίντου. Πρέπει να είναι δυνατόν για όλους μας να εκφραζόμαστε στις γλώσσες μας, αλλά όχι μόνο να εκφραζόμαστε, να ακούμε και όλα στις γλώσσες μας, γιατί είναι κουραστικό να παρακολουθούμε μία γλώσσα μέσω της διερμηνίας. Είμαι πεπισμένη ότι έχουν όλα τα δικαιώματα, ε, τα ίδια δικαιώματα όλοι οι ε, βουλευτές. Δεν μπορεί κάποιος ε, ο οποίος προέρχεται από χώρα με γλώσσα που έχει μεγαλύτερη διάδοση να έχει περισσότερα δικαιώματα και κάποιος άλλος που είναι από χώρα με, μικρότερη, με τις οποίες η γλώσσα έχει μικρότερη διάδοση να μην γίνεται εξίσου σεβαστός. Ευχαριστώ πολύ και συμφωνώ λέει ο Πρόεδρος και προχωρώ με τις ψηφοφορίες. We have two, Έχουμε δύο υπεράριθμους από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Όχι, κυρία Ρέγνερ, αποχωρεί. Έναν υπεράριθμο. So it seems to be okay. Please enter. Καλώς, τώρα είμαστε έτοιμοι. Παρακαλώ να ε, εισαγάγετε τις κάρτες για την ψηφοφορία όμως, όχι τις πιστοτικές, στο μηχάνημα. Πιστοτικές δεν γίνονται δεκτές. Η δική μου έκθεση πρώτα. Ηλεκτρονική δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας. Μοναδική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική παρακαλώ. Λείπει ακόμη ένας που δεν έχει ψηφίσει. Έγκρινεται. Μαστάλκα τώρα. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους κτλ. Τροπολογία υπαριθμών 13 υπέρ. Κατά αποχές και εγκρίνεται υπάρχει μόνο ένα κατά αποχές εγκρίνεται αριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 5 και 18 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε από το ΕΛΚ έχουμε έναν υπεράριθμο ας μην ψηφίσω εγώ λοιπόν Ωραία, τότε πάω εγώ να ψηφίσω. Γκρίνεται. Συμβαστική τρία, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 21 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά ας το επαληθεύσουμε εγκρίνεται 8, 22 και 23 παρακαλώ μαζί υπέρ κατά Θα ήθελα να σηκώνετε τα χέρια σας περισσότερο να τα βλέπω. Επαληθεύουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 9 και 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη σαν επαληθεύουμε Καλώς, συγκρίνεται. 25 όχι. Όχι. 26 ε, παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά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 ηλεκτρονικά το σύνολο της, ε, του σχεδίου. Και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μαστάλκα. Και έκθεση πάλι του κύριου Μαστάλκα. Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου. Ε, τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 παρακαλώ. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε 31 εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 30 συμβαστικέ συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά και να επαληθεύσουμε την 163 Απερίφθη. 37. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ. Κατά Ας επαληθεύσουμε την 168. Απρίφθη. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη αλλά ας επαληθεύσουμε είχε απορριφθεί 165 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 165 παρακαλώ Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Από χες εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Από χες απερίφθη. 171 υπέρ. Κατά Ας επαληθεύσουμε την 171 παρακαλώ. Αγκρίνατε. 172 υπέρ. Όχι, λάθος δικό μου. Σαράντα λοιπόν. 40 παρακαλώ υπέρ, κατά. Να κάνουμε μια παλήθευση για το 40. Απορρίπτεται. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Για τη 40. απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά να ελέγξουμε τη 43 παρακαλώ Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Δεν υπάρχουν πλειοψηφίες συνεχώς. Εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά εποχές πρέπει να ελέγξουμε και πάλι την 180 απορρίπτεται 181 υπέρ Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε ελεγχό. Ναι. Δικό μου λάθος εγκρίνεται. Πάμε στην 46 στην περίπτωση αυτή. 182, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 182 είμαστε. Ήμασταν μάλλον. Yes, 174 in favor. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ την 183 απορρίπτεται συμβαστική 15 υπέρ κατά εποχέ. Εγκρίνεται 48 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. Εποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται, έλα να ελέγξουμε. Εγκρίθηκε. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. Κατά εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 52 και 191 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά γκρίνετε εγκρίνεται το υπέρ κατά Συγγνώμη. 189 διορθώνει ο πρόεδρο. Υπέρ, κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 196 περ κατά εποχές απορρίπτεται να αλλάξουμε την 196 απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε τη συμβαστική 18 εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά εποχές μπορούμε να ελέγξουμε τη 2.11 Adopted. Εγκρίνεται. 2.12 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 215 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη 216. Εγκρίνεται. 2-18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την τροπολογία της κυρίας Χατάλα 2.20. Απορρίπτεται. Δύο υπέρ. Κατά. Εποχές, συγκρίνεται. 2,23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τη 25. My mistake. Εγκρίνεται. Δικό μου λάθος. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται η 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 231 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δύο υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Νομίζω εγκρίνεται. Ναι, εγκρίνεται. 2.34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.36 υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 2.37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.38 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται, 80 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Για να ελέγξουμε την 80. Απορρίπτεται. Με 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 240 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 248 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 250 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 2.51 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 255 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά 84. Διαθετήθηκε η 257. Επομένω πάμε στην 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 86 και 260 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται συγγνώμη 267 υπέρ κατά αποχές να ελέγξω 267 Εγκρίνεται 267. 269 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται 1 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται 88 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται 89 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά μπορούμε να ελέγξουμε τη 2 εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ όχι. Περνάμε στη συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά εποχή εγκρίνεται 96 υπέρ κατά εποχή εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά εποχή εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εποχή απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 114 Ελαφρώς υιοθετήθηκε. 113 υπέρ. Κατά. Θέλω να βλέπω τα χέρια σας. 113 υπέρ. Κατά. Μια απόπειρα ακόμη για την 113 υπέρ. The vote is rather long, you know, so forgive us. Uh, so we are at one. Λοιπόν, πάμε στα 115-116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε τη 16 Οπότε απορρίφθηκε. Λυπάμαι. Ζητώ συγγνώμη, εγκρίνεται η 16. Εκατόν 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά Εποχές. εγκρίνεται 19 υπέρ κατά Εποχές. εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά Εποχές. εγκρίνεται 127 υπέρ κατά Υιοθετήσαμε τη συμβαστική 7, επομένως πάμε στην 127, σωστά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 141 και 24 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Κυρία Χωτάλα πριν να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία πρέπει να πω ότι εξεπλάγει που αυτή η Επιτροπή θέλει να αυξήσει την αδιαφάνεια και τη μυστικότητα της ε, αξιολόγησης κινδύνου της αληθίδας τροφίμων αντί να κάνουμε αυτό που θέλει η Κομίσιο, να αυξήσουμε τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα. Και η μόνη μου ευκαιρία αυτό είναι να πάω να καταψηφίσουμε την πρόταση αυτή γιατί είναι σοκ αυτή η Επιτροπή να ζητήσει περισσότερη μυστικότητα και εμπιστευτικότητα, λιγότερη διαφάνεια και βιωσιμότητα. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Two more. No, okay, it's okay. And it has been adopted. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Μαστάλκα. May say something? Ε, θα ήθελα να πω κάτι. Με ενημέρωσαν ότι ο κύριος Μαστάλκα θα ήθελε να διαγραφεί το όνομά του από την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Θα το σημειώσουμε. Συνεχίζουμε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 εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ με ονομαστική κλίση Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Με. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Συγχαρητήρια στον κύριο Ράντεφ. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης με τη μορφή επιστολής για ε, την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης. Η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Η επόμενη ψηφοφορία θα γίνει και κλεισμένων των θυρών αργότερα. Τελείωσαν οι ψηφοφορίες λοιπόν προς το παρόν.

May Συνεχίζουμε με το σημείο 14. Αναφορά στην Επιτροπή για τον κανονισμό ΣΑΤΚΑΜ. Είμαι ο ίδιος εισηγητής. So, the fourth trilogue on the proposed SATCAP regulation was held at the Council. Λοιπόν, ο τέταρτος τριμερής διάλογος έλαβε χώρα αυτήν την Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου, Ήταν ο πρώτος τριμερής διάλογος κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας. Ο τριμερής διάλογος αυτός είχε στόχο την έβρεση μιας συνολικής πολιτικής συμφωνίας για τα κύρια πολιτικά ζητήματα, δηλαδή το ε, πεδίο εφαρμογή της επέκτασης της αρχής ε, για τη χώρα προέλευσης, το πεδίο εφαρμογή των αναμεταδόσεων και η τεχνική direct injection της άμεσης έγχυσης. Ενώ επετεύχθη ελάχιστη πρόοδος στους πρώτους τρεις διαλόγους, το Συμβούλιο πρότεινε να αλλάξει η μορφή του ε, μέσου, να γίνει δηλαδή από οδηγία, έτσι ώστε να βρεθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών ε, στο Συμβούλιο, κυρίως για το ζήτημα της άμεσης έγχυσης. Οι συζητήσεις κράτησαν μέχρι τα μεσάνυχτα ήταν πολύ επικοδομητικές. Σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος για την επέκταση της χώρας προέλευσης. Προτάθηκε αναδιατύπωση στο άρθρο 2, 2 και την αιτιολογική σκέψη 9β για να ληφθεί υπόψη η άποψη του Κοινοβουλίου ότι το πεδίο εφαρμογή ε, εκτό από το ραδιόφωνο και τι ε, ειδήσει και την επικαιρότητα θα πρέπει να καλύπτει μόνο προγράμματα τα οποία παράγονται εντό ε, των ραδιοτηλεπτικών οργανισμών και δεν θα συμπεριλαμβάνει συμπαραγωγέ. Για τις αναμεταδόσεις, η συμπερίληψη του ορισμού των managed environments, περιβάλλοντα υποδιαχείριση, συμφωνήθηκε προσωρινά και ένας ε, φορέας αναμετάδοσης θα παρέχει ασφαλή αναμετάδοση στους ε, εγκεκριμένους ε, βάσεις σύμβασης χρήστες. Συζητήθηκαν επίσης πιθανή αναθεώρηση στο άρθρο 12. Τώρα για την τεχνική της άμεσης έγχυσης επετεύχθη συμφωνία επί της αρχής για να συμπεριληφθούν διατάξεις έτσι ώστε να αλλάξει το μέσο και να γίνει οδηγία από κανονισμός. Η ακριβής διατύπωση των ε, διατάξεων αυτών εκρεμεί ακόμα. Θα συνεχίσουν τώρα οι εργασίες ε, σε λεπτομέρειες τεχνικού επίπεδου. Έχει προγραμματιστεί πέμπτος τριμερής διάλογος έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε οριστική συμφωνία και να ολοκληρωθεί ε, το θέμα στον τριμερή αυτό διάλογο. Να σημειωθεί ότι δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να ε, επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές που επιθυμούν να σχολιάσουν την ενημέρωση αυτή για τον τριμερή διάλογο. Δεν βλέπω να επιθυμεί κάποιο το λόγο. Το Συμβούλιο ή η Επιτροπή θέλουν το λόγο. Όχι. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν το σημείο αυτό και να συνεχίσουμε με το σημείο 15 υποβολή αναφορά στην Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Οδηγία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ο κύριος Φως έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συναντηθήκαμε λοιπόν στο πλαίσιο του πρώτου τριμερούς διαλόγου όπου συζητήσαμε αρχικά τις γενικές πολιτικές προτεραιότητες, έγινε ανταλλαγή απόψεων πάνω στα άρθρα 11 και 13, τα οποία χαρακτηρίσαμε πολύ σημαντικά πολιτικά. Αυτό δεν ήταν και δύσκολο, εξάλλου. Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για την εντολή των άρθρων 3 ε, έως 9α εκτός από το 14α για τη δίκαιη αποζημίωση και την ε, στοχευμένη συλλογή και εξόριξη δεδομένων. 14α δηλαδή ως 16α. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις ε, τεχνικού χαρακτήρα, θα θέλαμε κατά τη διάρκεια της Αυστριακή Προεδρία να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας έτσι ώστε να προετοιμαστούμε για ε, την συνέχεια, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τον, ε, το τεχνικό σκέλος του τριμερούς διαλόγου. Έχουμε ένα έγγραφο βάση το οποίο μπορούμε να ε, χτίσουμε. Θα χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση και στο πλαίσιο της ε, διδικασίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να το ε, χρησιμοποιήσουμε. Εδώ υπήρξε ένα ζήτημα ε, προσθήκης δύο άρθρων. Μετά συμφωνήσαμε για την ημερομηνία διεξαγωγής του τρίτου και του τέταρτου τριμερούς διαλόγου στις 26 Νοεμβρίου, τις 13 Δεκεμβρίου και στις 25 Οκτωβρίου. Αυτή η ημερομηνία ε, είναι λίγο αβέβαιη, δεν ε, γνωρίζουμε ακόμα αν θα καταφέρουμε να συναντηθούμε τότε, όμως ε, στο... πολύ σύντομα θα μάθουμε αν θα τα καταφέρουμε. Τρεις τριμερείς διάλογοι λοιπόν, τεχνικές συναντήσεις, νομίζω πως υπάρχει καλή βούληση Είμαστε θετικοί στο ότι θα τα καταφέρουμε. Στον επόμενο τριμερή διάλογο θα συζητηθούν τα άρθρα 3 έως 6, 14α έως 16α, 10α έως 12α και θα συζητηθεί ε, ξανά το άρθρο, τα άρθρα 13, 11 έως 13. Θα Φυσικά τα άρθρα 11 ως 13 δεν θα είναι τόσο εύκολο να ε, ολοκληρωθούν, αλλά με την πάραδο του χρόνου και με τους τριμερούς διαλόγου, διαλόγους θα καταφέρουμε να ε, τα ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν σχόλια από τους συναδέλφους. Όχι. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ το σημείο 15. Περνάμε στο σημείο 16. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης για τις διασυνοριακές αιτήσει επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λαιλατήθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις και πολέμους. Είμαι προσωπικά εγώ So I'm Με ενημερώνουν πως η έκθεση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα και αυτό μόλις χθες. Ας ληφθεί λοιπόν αυτό παρακαλώ υπόψη όταν θα εξετάσουμε τα χρονοδιαγράμματα. Το θέμα αυτό εστιάζει στις εκκρεμότητες και τις δυσκολίες ε, ιδιωτών για να ανακτήσουν έργα τέχνης και πολιτισμικά αγαθά τα οποία αποκτήθηκαν παρανόμως σε περίοδους πολέμου. Δεν υπάρχει φυστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία καλύπτει επαρκώς τις αιτήσει αποζημιώσεων από ιδιώτες. Μάλιστα, το διασυνοριακό στοιχείο είναι παρόν στις περισσότερες περιπτώσεις λαιλατήσεων, λαιλατημένης τέχνης από τη Συρία, από το Ιράκ, που πολίθηκαν στο Λονδίνο. Η έκθεσή μου συμφωνεί με την έκθεση για το νομικό πλαίσιο ελεύθερης κυκλοφορίας εντό αγαθών των οποίων η ιδιοκτησία αμφισβητείται εντός της ενιαίας αγοράς. Το Δεκέμβριο του 2003 η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέκρινε ένα ψήφισμα που καλεί τα κράτη-μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να εγκρίνουν μέτρα που θα διασφαλίζουν τη δημιουργία μηχανισμών ευνοϊκών προς την επιστροφή των αγαθών στους ε, νόμους δικαιούχους τους. Για περιπτώσεις λαϊλατημένης τέχνης. Την εποχή εκείνη είχαν μείνει εκκρεμότητες, δεν είχαν επιληθεί όλα τα ζητήματα και υπάρχει ο κίνδυνος, οι συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις να ε, προκαλέσουν περισσότερες δυσκολίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε, ε, το, το Κοινοβούλιο λοιπόν αποφάσισε να καταρτήσει έκθεση πρωτοβουλίας. εξετάζεται ε, η δυνατότητα χρήσης μηχανισμού επίλυσης διαφορών, ο οποίος ενδεχομένως είναι καταλληλότερος και προσφέρει λύσεις πιο ευέλικτες που μπορούν να προσαρμοστούν στην κάθε περίπτωση λύσεις όχι αυστηρές που ευνοούν φιλική επίλυση των διαφορών. Επίσης, εξετάζεται η δυνατότητα ε, δημιουργίας ε, κοινών καταλόγων που θα συλλέγουν δεδομένα για τις περιπτώσεις ε, αγαθών και έργων τέχνης που είναι αποτέλεσμα λαϊλασίας. Θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε όχι μόνο με τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στο παρελθόν, αλλά και με την πρόληψη και επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν ε, στο μέλλον ως αποτέλεσμα ένοπλων ε, συγκρούσεων που θα οδηγήσουν σε λαϊλασίες ή σε αναγκαστική πώληση των αγαθών αυτών. Θα ήθελε κάποιο μέλος το λόγο? Όχι. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο? Όχι. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 5 Νοεμβρίου. Ψηφοφορία στις 20 Νοεμβρίου στην Επιτροπή. Αυτά λοιπόν για το σημείο 16. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρωινής μας συνεδρίασης. Καλή όρεξη λοιπόν. Θα τα πούμε στις 2.30 το απόγευμα.